the vote. Okay. Good morning. Καλημέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. We thank you for your cooperation, those in the hall. Try to concentrate, be seated. Παρακαλώ προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε οι όρθιοι να καθίσουν. Καλημέρα σας. Σήμερα το πρωί συνεδριάζει ολόκληρη τη μέρα μάλλον η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η συνεδρίαση των συντονιστών που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 11.30 αναβάλλεται για τις 17 Οκτωβρίου. Έχουμε και άλλες μικροαλλαγές. Θα, στα, σας τις αναφέρω γύρω στις 10 ε, και 4, οπότε θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ανακοινώσει του Πρόεδρο τώρα. Καταρχήν σας υποβάλλω προς έγκριση τις συστάσεις των συντονιστών, οι οποίες είναι εξής. Καταρχήν, ο συνάδελφος Σαλβατόρη Γιακολίνο ορίστηκε εισηγητής της πρότασης για την δημιουργία του γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Δεύτερον, ο κ. Αξελβός ορίστηκε εισηγητής της πρότασης κανονισμού για την αναθεώρηση του κανονισμού για τη δομή του Eurojust. Τρίτον, ο συνάδελφος Γιάτσεκ Προτασέβιτς ορίστηκε εισηγητής ε, στον κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις νέες ε, ψυχοδραστικές ουσίες. Και κατόπιν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, εγκρίνονται αυτές οι στάσεις των συντονιστών. Και επίσης η ψηφοφορία για την προστασία των δεδομένων θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 και κατά πάσα πιθανότητα και στις 24 Οκτωβρίου από 10 με 12 στο Στρασβούργο. Επίσης έχουμε και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων μας και μάλιστα έχουμε και την μέχρι τα τέλη του έτους την έρευνα της Επιτροπής όπως έχει εγκριθεί από τους συντονιστές. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, να περάσουμε στην έγκριση των πρακτικών των τριών τελευταίων συνεδριάσεων του Οκτωβρίου, Απριλίου και Μαΐου. Αγκρίνουμε τα πρακτικά αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και περνάμε στο σημείο 4 την τρέχουσα κατάσταση των ενεξελίξη διοργανικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Έχουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Μέλο, που θα μας ενημερώσει για Ποια έκθεση μιλάμε? Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνη. Έχουμε εδώ, είπα τον εισηγητή μας, ε, για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Έρευνας, τον κύριο Μέλο, που θα μας ενημερώσει για την πρόταση για τις εξελίξεις των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Δεν έχω να σας αναφέρω πολλά σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση. Θα ήθελα απλώς να πω ότι στη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας σημειώσαμε εντυπωσιακές προόδους σε πολλά άρθρα. Έχουμε περάσει τώρα στη Λιθουανική Προεδρία. Οπότε θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις για συγκεκριμένα τμήματα της έκθεσης και ελπίζω στις αρχές του επόμενου έτους να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση και να ψηφίσουμε. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Άλλα σχόλια δεν υπάρχουν. Ακούσαμε λοιπόν την ενημέρωση από τον εισηγητή για τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης. Δεν υπάρχουν άλλες εξελίξεις στις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγετής μας είναι ο κύριος Λουί Μισελ που, συνέταξε την ετήσια, που σχολιάζει την ετήσια έκθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμεί είμαστε η αρμόδια επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των ε, δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στην Ένωση. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν το σχέδιο έκθεσης του κύριος ε, Λουί Μισελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να θυμίσω απλά ότι η δομή της έκθεσης αφιερώνεται σε μια, ένα πρώτο τμήμα που αφορά τους ε, θεσμικούς οργανισμούς που έχουν αναλάβει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά ακολουθεί ένα δεύτερο τμήμα που εξετάζει τα συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ακολουθώντας τη δομή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα κεφάλαια για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ηθαγένεια και την δικαιοσύνη. Όσον αφορά το θεσμικό τμήμα, όπως ξέρετε, έχουμε γνωρίσει, γνωρίσει κρίσεις ε, θεσμικού τύπου και συνταγματικού τύπου εξαιρετικά σημαντικές σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπήρχε η ε, έξωση των ε, Ρωμά στην Γαλλία, η κρίση στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία και μάλιστα το κοινό ε, παρονομαστής είναι η παραβίαση ή η υποψία παραβίασης σύμφωνα με το άρθρο 2 ε, της Συνθήκης περί Ευρωπαϊκής Ένωσης Τις τελευταία, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή συζήτηση όσον αφορά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και μέσω αυτής της συνθήκης ή που θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω τροποποιήσεων των συνθήκων ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο και συγκεκριμένα μέσω ενός νέου μηχανισμού. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά εδώ και χρόνια μια πολιτική και μέσα πιο ε, καθοριστικά για τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο εργασίε που έχω υποβάλει στην Επιτροπή συμπεριλαμβάνουν τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, αλλά και προτάσει για ενίσχυση τη πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων με, σύμφωνα με τι ισχύουσε συνθήκε, αλλά και εν ώψη τροποποιήσεων αυτών. Η κυρία Ρέντινγκ έδωσε κάποιες υποδείξεις, κάποιες ενδείξεις μάλλον για τις προθέσεις της Κομισιόν στη διάρκεια της παρέμβασή της στην πρόσφατη διάσκεψη του Κέντρου για την ε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Πολιτικές Σπουδές, Μελέτες και εστίασε την προσοχή στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διάφορα στοιχεία του άρθρου 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε να χρησιμοποιηθούν ε, ε, ε, επιστολές στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 7 της Συνθήκης, που αντιστοιχούν στην τυποποίηση μιας πρακτικής που η Κομισιόν έχει χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, με την Ουγγαρία. Προτείνει επίσης να προβλεφθεί μια σειρά ε, τροπολογιών στις συνθήκες που είναι θετικές αλλά εμπεριέχουν ένα κίνδυνο την ε, παραπομπή στις ελληνικές καλένδες του μηχανισμού αυτού του νέου ε, μηχανισμού και της εφαρμογής του. Εμείς συμμεριζόμαστε τους στόχους ενίσχυσης του μηχανισμού ε, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, θεωρούμε πως έχουμε διαφορετικό όραμα σε σχέση με το τι μπορεί ήδη να κάνει η Κομισιόν σύμφωνα με τις ισχύουσε συνθήκες και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αυτών των ρυθμίσεων. Θεωρώ επίσης πως δεν πρέπει μόνο να εργαστούμε για να εγγυηθούμε το κράτος δικαίου, αλλά και για να εγγυηθούμε την εφαρμογή του άρθρου 2 της συνθήκης στο σύνολό του, δηλαδή δημοκρατία, κράτος δικαίου, ε, θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα και μειονότητες για να μπορέσουμε πλήρως να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της, ε, της, ε, των συνθηκών θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε τη μεταγραφή των, του Ευρωπαϊκού Δικαίου που αγγίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προβλέψουμε συγκεκριμένες πολιτικές υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινών αξιών. Να συνεργαζόμαστε με πιο συστηματικό τρόπο με το Συμβούλιο της Ευρώπης και, άλλα και άλλους διεθνείς θεσμούς που ασχολούνται με το ίδιο θέμα και να φτιάξουμε ένα νέο μηχανισμό που στόχο θα έχει <coughs> την εγγύηση του σεβασμού, της πρόθεσης και την προστασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να, μπορεί η Κομισιόν, αν επιθυμεί, να υιοθετήσει μια απόφαση, όπως το έκανε για την παρακολούθηση στο πλαίσιο των κρατών μελών, ώστε να φτιαχτεί ένας τέτοιος νέος μηχανισμός. Ε, δεν χρειάζεται τροποποίηση των συνθηκών, για παράδειγμα, για να οριστούν δείκτες για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της παρακολούθησης της κατάστασης εντός της Ένωσης και στα κράτη-μέλη για να γίνουν αντικειμενικές μελέτες για να φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό site για την εφαρμογή του άρθρου 2 της συνθήκης και για να αναπτύξουμε και να νομοθετήσουμε για ένα σύνολο κυρώσεων. Επίσης για τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Όλα αυτά ήδη μπορεί να τα κάνει η Κομισιόν αν το επιθυμεί σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες. Πρέπει δηλαδή κατ' να εφαρμοστούν όλα τα μέσα που αυτή τη στιγμή προβλέπονται από τη συνθήκη και να προετοιμάσει και τροποποιήσει για τη συνθήκη και όπου αυτό χρειάζεται. Για το τμήμα που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως σας έλεγα, ακολούθησα τη δομή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, εξέτασα και τα έγγραφα των πιο σημαντικών ΜΚΟ για να διαπιστώσω τις πιο ανησυχητικές παραβάσεις στα κράτη-μέλη και στην Ένωση, όπως και σε αυτές που είναι οι πιο συχνές στα, εκθέσει των ΜΚΟ. Εξαιρετικά πολλές περιπτώσεις όσον αφορά την παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πολλές, πολλά περιστατικά στην Ένωση και σε ορισμένα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μειονότητες, τους ετούντες άσυλο, τους μετανάστες, τα άτομα που είναι ύποπτα για σύνδεση με την τρομοκρατία ή αυτούς που στερούνται της ελευθερίας τους. Θα πρέπει να σεβαστούμε απόλυτα την απαγόρευση βασανιστήριων και των απάνθρωπων, της απάνθρωπης μεταχείρισης ε, γιατί όλα αυτά βασίζονται στην, στο σεβασμό των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει αυστηρά να τηρούνται είτε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είτε στο πλαίσιο τη διεθνού συνεργασία. το δικαίωμα στην προστασία και το σεβασμό της, της ιδιωτικής ζωής είναι μια ουσιαστική αξία όπως και η ελευθερία ενημέρωσης και έκφρασης των ΜΜΕ που είναι πολύ σημαντική σε μια δημοκρατία. Εξαιρετικά πολλές περιπτώσεις παραβίασης του δικαίωματος ασύλου ε, και, και παραβιάσεις κατά τη διάρκεια έκδοσης ε, ε, μεταναστών συμβαίνουν δυστυχώς ακόμη. Και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τον αγώνα της κατά των διακρίσεων να υιοθετήσει την οδηγία που σχετίζεται με την αρχή της ισότητας της μεταχείρισης των ανθρώπων χωρίς διάκριση θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ε, ηλικία κτλ. Η κατάσταση των Ρωμά παραμένει πολύ ανησυχητική. Πρέπει επισήμω να καταδικάσουμε κάθε τύπου βία ρατσιστική κατά μειονοτήτων ε, ή μεταναστών και λυπούμεθα για την έλλειψη δράσης από πλευράς των αρχών οι πολιτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν τους Ρωμά ως αποδιοπομπαίους τράγους όπως είδαμε και την τελευταία περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία. Η κρίση πολύ συχνά πλήττει τις πιο φτωχές ε, ε, ομάδες των πληθυσμών μας και γι' αυτό θα πρέπει να τους δοθεί πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Το δικαίωμα στην ελευθερία ε, κυκλοφορίας είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη και τα πιο ορατά που έχουν οι πολίτες της Ένωσης. Μπορούμε ε, να θα πρέπει να αναχαιτήσουμε κάθε απόπειρα που στόχο έχει να, να τρέψει αυτό το, το κεκτημένο. Θα πρέπει να είναι η ε, Κομισιόν και τα κράτη δίκαια, ισότιμα, για να δουλέψουν υπέρ του κράτους δικαίου. Δεν μπορεί φυσικά να ισχύσει ούτε να γίνει ανεκτή καμιά ατιμορρησία συντομία, να, λοιπόν, σας ανέφερα τα διάφορα σημεία της εκθεσής μου. Είναι πραγματικά ε, δύσκολο γιατί θα μπορούσα να αναπτύξω περισσότερο κάποιες πτυχές όπως τα δικαιώματα των παιδιών, τη θέση των αναπήρων στην κοινωνία, την κατάσταση των μειονοτήτων και τα κοινωνικά δικαιώματα. Αλλά αυτή τη στιγμή οι κανόνες παρουσίασης των εκθέσεων πρωτοβουλία δεν μας επιτρέπουν δυστυχώς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Προβλέπω ήδη να καταθέσω μια σειρά τροπολογιών ώστε να μπορέσω να αναπτύξω και να εντάξω στοιχεία τα οποία ξέφυγαν ή έμειναν στην άκρη για την ώρα. Θα ε, φτιάξω και μια σειρά προτάσεων για τους σκιώδεις εισηγητές που μπορούν να τις υπογράψουν αν το επιθυμούν. Θεωρώ επίσης πως για να εμβαθύνουμε στην ε, συζήτηση πρέπει να συζητήσουμε για την πιθανή δημιουργία μιας επιτροπής της Κοπεχάγης και να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα δημιουργίας μιας τέτοιας επιτροπής και για να συνεχιστεί ο προβληματισμός μας για αυτά τα θέματα που πρέπει να μείνουν στην καρδιά της δράσης μας. Διοργανώνονται στις 5 Νοεμβρίου, ε, διοργανώνεται ακρόαση και σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά. Η προθεσμία γιών είναι η 11η Νοεμβρίου, πράγμα που μας αφήνει χρόνο για να το σκεφτούμε και για να ακούσουμε και τις ακροάσεις πριν να υποβάλουμε ατροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Λου Μισελ. Το λόγο κύριος Μέλο. Αγαπητά μέλη, εκ μέρους του ΕΛΚ και εκ μέρους της και ηγήτριας κυρίας Μπάουερ, θα ήθελα να σα ε, αναφέρω την άποψη τη πολιτική μου ομάδα. Καταρχά, να σα πω ότι το ΕΛΚ δίνει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση και βελτίωση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, στι παραγράφου 2 και 7 τα σημεία που αναφέρονται απέχουν πολύ από την πραγματικότητα για την προστασία των πολιτών. Καταρχά, δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτύξει ένα αναπτυγμένο σύστημα προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, είτε νομικά είτε θεσμικά η πρόταση του εισηγητή επιφέρουν μεγάλο κίνδυνο ε, της προστασίας των πολιτών και αυτό πρέπει να αποφευθεί κατά, οπωσδήποτε. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σύστημα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και να σας θυμίσω ότι μετά από σύσταση του Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνέστησε ένα δίκτυο πυρογνωμόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο ανέλαβε να συντάξει ένα σχέδιο έκθεσης κατόπιν πρόσκλησης των κρατών μελών. Η δημιουργία ενός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, έλαβε χώρα το 2003 και ο Επίτροπος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίστηκε το 2009. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτησε ένα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και την ηθαγένεια από το 2007 μέχρι το 2013, το οποίο συζητούμε και τώρα. Να τονίσω επίσης ότι η Σύμβαση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα έχει, είναι νομικά θεσμευτική για τις συνθήκες και τώρα είναι βασικό συστατικό στοιχείο της νομικής μας ε, βάσης. Αναφέρεται στις βασικές αρχές του κράτους δικαίου και καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και πέρα από αυτό. Σύντομα θα ακολουθήσει μια αξιολόγηση εν ώψη της ε, Σύμβασης ε, για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα για την ε, σωστή λειτουργία του συστήματος και πρέπει να αποφύγουμε όπως και δίποτε μια πολιτικοποίηση ε, για των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα επιχειρήματα που θέτει ο εισηγητής για τη δημιουργία νέων οργάνων πέρα από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιφέρει κίνδυνο αυτής ακριβώς της πολιτικοποίησης. Το σύστημα πρέπει να παραμείνει ε, πέρα και εκτός από κάθε ε, πολιτική βούληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο παραμένουν πολιτικά όργανα, γι' αυτό λοιπόν η προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων παραμένει νομική αρμοδιότητα των ε, θεσμικών οργάνων όπως ε, το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δικαστήριο των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Και αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 της συνθήκης. Η αναφορά σε αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνη διότι υπάρχει ο κίνδυνος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, μην είναι πλέον αμερόληπτο όσον αφορά την ε, προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κλέης επίσης ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. πιστεύω πως αυτή η έκθεση είναι μια χαμένη ευκαιρία για εμάς. Εδώ υπάρχει ένας ε, μακρύς κατάλογος θεμάτων τα οποία μας δείχνουν ότι, τα, ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη η έκθεση δεν περιέχει και κάτι καινούριο, δεν φύγει ε, νέα ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην παράγραφο 15, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι εκφράζεται η ανησυχία για διάφορες παραβιάσεις ε, ασύλου και γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις ε, που δεν τηρούνται από ορισμένα κράτη-μέλη. Αναφέρεται ο κίνδυνος που διατρέχει η ζωή ανθρώπων που προσπαθούν να ε, περάσουν τα εξωτερικά σύνορα. Αυτό μου φαίνεται πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά, αλλά και ορισμένοι συναδελφοί από αυτήν την Επιτροπή, ήμασταν σε μια αποστολή στην Ισπανία, πήγαμε στο Γιβραλτάρ και εκεί είδαμε πως η αστυνομία, η Frontex και οι συνοριοφύλακες κάνουν καλά τη δουλειά τους, την παίρνουν στα σοβαρά. σχετικά με όσους προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Γιβραλτάρ. Και πιστεύω πως το ίδιο γίνεται και σε άλλες περιοχές που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Το ίδιο και με τις ελιμενικές αρχές. Αυτοί, αυτές οι, αυτοί άνθρωποι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και δεν πιστεύω πως αυτή η έκθεση είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναφερθούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ε, κατηγορίες για ανθρώπους οι οποίοι πιστεύω πως κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται θύματα, αλλά κανείς δεν έχει πει ότι εκείνοι οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη του εαυτού τους. Και πάλι βρίσκω πως αυτή η έκθεση δεν εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που έχει. Η παράγραφος 18 αναφέρει ότι για μία ακόμη φορά ε, ο ρατσισμός είναι καταδικαστέος, ιδιαίτερα ο ρατσισμός προς τους ε, μετανάστες, αλλά γιατί δεν μιλάμε και για τον ρατσισμό που προέρχεται από τους μετανάστες σε πολλές ε, γαλλικές ε, πόλεις υπάρχει ρατσισμός από τους μετανάστες προς τον ε, τόπιο πληθυσμό και ίσως ο εισηγητής θα μπορούσε να είχε αφιερώσει κάποιο χώρο στην έκθεση για αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας τον Λουί Μισελ για την έκθεση του που πραγματοποιεί σημαντικά βήματα στο μονοπάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κατάστασης δικαίου, των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα εδώ και χρόνια ενεργοποιείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά και η έκθεση συνεχίζει την ε, κρατούσα άποψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια ολόκληρα. Ε, στα πλαίσια της συζήτησης για το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, ο χάρτης αυτός, στην παρούσα μορφή, δεν εφαρμόζεται στην εσωτερική ενόμη τάξη των κρατών μελών, εκτός ε, και αν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και δυστυχώς η σημερινή κατάσταση υστερεί σε σχέση με τις φιλοδοξίες και το ζητούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχουμε ακόμη και στα κράτη-μέλη παραβιάσεις ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Και μάλιστα αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να εκφράζουμε ωραία και μεγαλεπίβολα λόγια το χάρτη θεμελιού δικαιωμάτων, ωραίο άρθρο 2 στην ε, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να έχουμε εμπράκτος παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό των κρατών μελών. Υπάρχει ασυνέπεια και μερικές φορές αυτή η παραβίαση παραμένει τιμόρυτη. Και γι' αυτό χρειάζεται μια ενίσχυση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ένωμης τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και συζητούμε για το άρθρο 2 και την συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε αυτή ήταν η γνώμη του ΕΛΚ και γνωρίζω βέβαια ο κύριος Μέλο ουσιαστικά αναπληρώνει εδώ την κυρία Ντιτ Πάουερ, της και αλλά η θέση του ΕΛΚ συνιστά παλινδρόμηση σε σχέση με την ε, παραδοσιακή στάση του ΕΛΚ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόσφατα μάλιστα η Επίτροπος Ρέντινγκ τάχθηκε υπέρ της διαγραφής του άρθρου 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που περιορίζει την ε, εφαρμογή ακριβώς του χάρτη. Εδώ εκφράζω και την προσωπική μου γνώμη, αλλά και την άποψη της ομάδας ε, και τη θέση της κοιόδης ηγετρίας κυρίας Λούνατσεκ. Η θέση λοιπόν της κοιόδης ηγετρίας ε, και της ομάδας ε, είναι ότι για να γίνει αποτελεσματική έκθεση θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα παράρτημα με λεπτομεριακή απαρίθμηση αναχώρα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα αυτό το στόχο θα έχουν και οι τροπολογίες που θα υποβάλουμε ως ομάδα. Και μέχρι τις 11 Νοεμβρίου θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με τον εισηγητή για να έχουμε αναφορά αναχώρα, όπως απαιτούμε εδώ και χρόνια. Θα πρέπει αυτή η λεπτομεριακή ενημέρωση αναχώρα για τις παραβιάσεις που γίνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επισυναυθεί στην ετήσια έκθεση και να συνοδεύει τα θεσμικά θέματα που επίσης είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει η συζήτηση για αυτά να διεκπαιρεωθεί αλλά να έχουμε και μια γενική επισκόπηση της κατάστασης στην Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελευταίο θέμα, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε την διαδικασία προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωση στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βέβαια, θα πρέπει να αποφύγουμε ταυτόχρονα και εδώ θα ήθελα να ακούσω το σχολιασμό του εισηγητή. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφύγουμε ένα είδο καταμερισμού των εργασιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γιατί υπάρχει ο πειρασμό αυτός μερικές φορές. Δηλαδή, να διαχωριστούν τα καθήκοντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αρμόδια μόνο για την εσωτερική αγορά και κάποιους μηχανισμούς συνεργασίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης να ε, είναι αρμόδιο για την προστασία του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών. Αυτός ο επιμερισμός των εργασιών θα αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό την ίδια την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πολίτες. Ταυτόχρονα θα αποδυναμώσει και το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί έτσι θα αφήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης μοναδικό αρμόδιο για το θέμα της, του κράτους δικαίου σε, στην επικράτεια 40 χωρών. Ένα τεράστιο πεδίο δηλαδή, που θα είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί. Γιατί έχουμε πολύ συχνά καταγγελίες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες μέλη. Οπότε το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πολύ μεγαλύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων, γιατί έχει πολύ περισσότερα μέλη σε σχέση με το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το άρθρο 2 και 3 της ε, Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας λένε ότι πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών και αρχών. Σεβασμός αξιοπρέπειας, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις αξίες, ελευθερία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και το καθεξής. Και στο 3.1 αναφέρεται ότι η πρωταρχική υποχρέωση της Ένωσης και η καθήκον της είναι η προώθηση αυτών των αξιών. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αναθέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή την προάσπιση των αξιών, ουσιαστικά παραβιάζει βασική της αρμοδιότητα που κατοχυρώνεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ανταποκρίνεται στο καθήκον της απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, η Επιτροπή της Κοπεχάγης θα πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία φυσικά με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα πρέπει να αποφεύγονται επικαλύψεις με την Επιτροπή της Βενετίας και θα πρέπει διμερώς να συνεχίσουμε τις συνεννοήσεις μετά από επαφές και διαβουλεύσεις που είχαμε με την Επιτροπή της Βενετίας στα πλαίσια από συζητήσεων για πολλές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αντιδράση Επιτροπής της ε, Βενετίας ό,τι αφορά την ε, δημιουργία της Επιτροπής Κοπεχάγης είναι, οι αντιδράσεις είναι πολύ θετικές γιατί και τα μέλη της Επιτροπής Βενετίας θεωρούν ότι μπορούμε να έχουμε μια, ένα πιο ε, αυστηρό όργανο. δεν υπάρχει καμία αντίφαση στην συμμετοχή και του Συμβουλίου της Ευρώπης στο έργο της Επιτροπής Κοπεχάγης. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Φυσικά θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, αλλά όπως είπε και ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ, μεταφέροντας τα σχόλια της και οδησηγήτρης κυρίας Μπάουερ, εμείς θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα πολιτικό θεσμικό όργανο το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα μετά τις επόμενες ευρωεκλογέ. Οπότε, η δημιουργία μη πολιτικών αρχών για την παρακολούθηση της ε, κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό βήμα που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και ε, θα είμαστε απόλυτα συνεργάσιμοι με τον εισηγητή. Κυρία Τσίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σταβάρες. Να πω όμως ε, ότι καταρχάς πιστεύω πως δεν θα ανταποκριθούμε στις ε, απαιτήσει των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν ε, συνεχίσουμε να θεωρούμε με τόσο περιορισμένο τρόπο τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτα να υπάρχει οδηγία και μετά να βλέπουμε δηλαδή αν τηρείται η οδηγία πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν από εμάς να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα συνέχεια, ανα πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πολιτικά, διότι πάντα παρατηρούμε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όταν ασκούμε κριτική σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό το κάνουμε στα πλαίσια της δημοκρατικής μας κουλτούρας, έχουμε και εμείς υποχρέωση να ασκούμε κριτική απέναντι στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καθήκον μας να προστατεύουμε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ έχουμε καθήκον να κάνουμε καλή δουλειά. Εάν δούμε το θέμα αυτό μόνο νομικά, δεν θα, δεν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη θεώρηση. Φυσικά και είναι πολιτικό το θέμα. Η πολιτική όμως συζήτηση για την τήρηση των ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και εμείς ως πολιτική ομάδα θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό μέσο που θα κάνει εξίσου αποτελεσματική αξιολόγηση αλλά και θα ασκήσουμε κριτική για όσα ε, σημεία πρέπει να βελτιωθούν και να αλλάξουν. Ο κύριος Στίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, μιλώντας για δικαιώματα, ε, δυστυχώς ε, δεν μπορώ σήμερα να μιλήσω κροατικά, δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Και ελπίζω την επόμενη φορά να αλλάξει αυτό. Θα μιλήσω λοιπόν αγγλικά μιλώντας για θεμελιώδη δικαιώματα και για την προώθηση των ε, ευρωπαϊκών αξιών, πιστεύω πως ε, για να είναι πιο ε, συνεκτική η έκθεση πρέπει να υπάρχει μια έκκληση στα κράτη-μέλη. Να συμμορφώνονται με όλα τα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι όταν μιλάμε για θεμελιών δικαιώματα, μιλάμε για ελευθερία, μιλάμε για το να καταδικάζουμε όλα τα καθεστώτα που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009 που καταδικάζει όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα, όχι μόνο κυβερνήσεις. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι ορισμένες χώρες στην κεντρική Ευρώπη έχουν συμμορφωθεί απόλυτα με αυτό το ψήφισμα, ορισμένες όμως όχι. Όπως και η κυρία Ζήπελη είπε, το θέμα δεν είναι μονονομικό, είναι και πολιτικό. Και υπάρχουν δύο επιμέρους ε, ζητήματα. Το πρώτο είναι η προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ζητήματα ως αφορμή για ε, πολιτική συζήτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες προσπάθειες χρήσης νομικών μέσων για να πλοκάρουμε οποιαδήποτε προσπάθεια συμφιλίωσης και να δημιουργηθεί ένα κλίμα εντελώς φιλόξενο για οποιοδήποτε απολυταρχικό καθεστώς στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη συγκεκριμένα. Πιστεύω λοιπόν πως για να είναι πιο περιεκτική η έκθεση πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτέ οι απόψει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πλένκοβικ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να συγχαρώ καταρχάς τον εισηγητή για τη δουλειά του σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και προερχόμενος από ένα νέο κράτος μέλος, είχαμε κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων προσχώρησης ε, δώσει πολύ μεγάλη σημασία στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Και κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων, εμείς ως Κροατία συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντικά είναι τα κεφάλαια για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτός ο τομέας ήταν ο πιο ευαίσθητος ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το πόση δύναμη έχει. και μαζί και όλας και το κεκτημένο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και σε μελλοντικέ διαπραγματεύσει προσχώρηση, η εμπειρία μα έδειξε πω αυτό το κεφάλαιο θα είναι ακόμα σημαντικότερο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τι ε, διαπραγματεύσει προσχώρηση με το Μαυροβούνιο, αλλά και με άλλε χώρε στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι πολύ, ε, πολύ σημαντική αναφορά στο άρθρο 2 στην έκθεση και αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε απόλυτα. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη δημιουργία νέων μηχανισμών οι οποίοι θα επιτηρούν και θα επιβλέπουν το ρόλο των θεσμικών οργάνων στην ε, προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Να τονίσω εμείς επίσης πως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Κροατία όταν το 2012 δεν ήταν ακόμα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε συμμετέχει στην ε, έκθεση και στην ανάλυση όλων των ε, επιμέρους ε, σημείων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και πιστεύω πως η χώρα μου ήταν, έδειξε πως ήταν πανέτοιμη να σεβαστεί απόλυτα όλα τα, τις πτυχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωραία. Ας ακούσουμε τώρα την ε, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν ε, επαναφέρομαι τον εισηγητή στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδραιώνεται σε σημαντικές κοινέ αξίες. Δεν πρέπει να τις παίρνουμε δεδομένες. Θα πρέπει να δείξουμε στους ε, πολίτες μας ότι ε, έχουμε δυνατότητα αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης αυτών των αξιών. Αυτό μάλιστα επισήμανε και ο πρόεδρος Μπαρόζο στην ε, έκθεση που έκανε για την κατάσταση της Ένωσης φέτος. Γιατί υπάρχουν προκλήσεις ε, στο κράτος δικαίου, ακόμη και εντός των κρατών μελών. Τόνισε για την ανάγκη γεφύρωσης της πολιτικής πυθούς και στις στοχευμένες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων αφενός και αφετέρου της χρήση του άρθρου 7 της συνθήκης, δηλαδή διακοπή ή μάλλον προσωρινή αναστολή των δικαιωμάτων του κράτους μέλους. Και μάλιστα εξήγηλε και την υποβολή όσον είπα μιας ανακοίνωσης ε, για το θέμα αυτό. Η εμπειρία μας έχει δείξει πόσο χρήσιμη είναι η θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ανεξάρτητο διοικητή. Και μάλιστα έχουμε προτάσεις για το μηχανισμό κράτους δικαίου, όπως ε, θα δείτε και στην ανακοίνωση που ετοιμάζουμε. Οι βασικές ε, αρχές είναι ότι ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει ε, σοβαρό συστημικό κίνδυνο στο κράτος δικαίου και ότι θα πρέπει να υπάρχουν προηγουμένως σημαντικοί συγκριτικοί κανόνες που θα εξασφαλίσουν ισοτιμία των κρατών μελών και μόνο έτσι θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Η ισοτιμία είναι πολύ σημαντική ε, στην περίπτωση αυτή. Δεν επιτρέπονται διπλά μέτρα και σταθμά. Πρόθεσή μας δεν είναι σε καμία περίπτωση να έχουμε επικάλυψη με υπάρχοντες μηχανισμούς, ε, ούτε με το Σύμβουλο της Ευρώπης, αλλά να εφοδιαστούμε με κάποιους μηχανισμούς αντίδρασης σε περίπτωση που διακυβεύεται το κράτος δικαίου σε μία περισσότερες χώρες μέλη. Θα πρέπει επίση να ξεκινήσουμε διάλογο και διαβουλεύσεις με όλους του ενδιαφερομένους και στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσει τον Νοέμβριο το Φόρουμ τη Δικαιοσύνης, μια διάσκεψη για το ρόλο της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το κράτος δικαίου και ο σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων θα αποτελέσουν το επίκεντρο τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν και ο εκπρόσωπος της Λιθουανικής Προεδρίας θα ήθελε να πει δυο λόγια πριν ακούσουμε και πάλι τον εισηγητή. Ενδιαφέρεται το Συμβούλιο. Είδε μη να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Λουί για να ολοκληρώσει. Δεν έχω την αίσθηση θα ολοκληρώσω. Απλώς θα απαντήσω εν συντομία στους συναδέλφους. Ομολογώ ότι έμεινα εμβρόντιτος από την ε, παρουσίαση του αξιότιμου συναδέλφου Μέλο, που λέει ότι με την έκθεση αυτή διατρέχουμε τον κίνδυνο πολιτικοποίησης του θέματος. Μα κύριε Μέλο, ακριβώς το αντίθετο κάνω με την έκθεσή μου. Γιατί στην έκθεσή μου προτείνω μια αντικειμενική και σαφή διαδικασία με, τη βάση, με βάση δικτών που σε καμία περίπτωση δεν είναι πολιτική γιατί σήμερα δεν είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση και μάλιστα από το ύφος και τον τόνο της ε, εισήγησή σας ε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ακριβώς ε, έκφραση της πολιτικοποίησης που ήδη επικρατεί στην συζήτηση αυτή. Γιατί δεν είναι καλό να εθελοτυφλούμε ιδιαίτερα ευρωβουλευτές, γιατί εθελοτυφλία είναι να πούμε ότι ότι συνδέουμε τα προβλήματα της Ευρώπης, ε, ε, τα προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θέματα στα κράτη-μέλη, τι να σας πω. Εγώ διαβάζω τις λεπτομεριακές εκθέσεις και διαπιστώνω ότι σε όλες τις χώρες μέλη, ακόμη και στη δική μου πατρίδα, έχουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κόσμος δεν είναι ρόδινος, δεν είναι τέλειος. Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δράσεις μας. Μου είπατε ότι δεν είμαι, δεν είμαι ρεαλιστής. Μα νομίζω ότι είμαι υπερβολικά ρεαλιστής. Το Συμβούλιο ζήτησε ένα νέο μηχανισμό. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην με κατηγορείτε λοιπόν για ουτοπία ή έλλειψη ρεαλισμού. Διαπιστώνεται ανάγκη ενίσχυση του οπλοστασίου μας, του ρυθμιστικού, για να διαθετήσουμε μια σειρά προβλημάτων. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την έκθεση του ΕΛΚ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και εσείς ενδιαφέρεστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε καμία περίπτωση δεν αφισβητώ την προσήλωσή σας ε, ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αλλά παρακαλώ διευρύνετε λίγο τον ορίζοντα το, του προβληματισμού σας και σε, σε καμία περίπτωση να μην κάνετε δίκη προθέσεων για απόπειρα πολιτικοποίησης του θέματος αυτού. Επουδενή δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Βέβαια, είμαι ελεύθερος συζητητής να συντάξω την έκθεσή μου και θα υποβάλω και ανεπίσημη έκθεση για όλες τις περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναχώρα. Ξέρω ότι ενοχλεί αυτό το θέμα και φυσικά δεν θα περιληφθεί στην επίσημη έκθεση γιατί πολλοί είναι κατά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα με εμποδίσετε ασκώντας την ελευθερία έκφρασής μου να επισημάνω και να καταγγείλω σοβαρές και κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. γιατί ε, τώρα και άλλες διαρρώσεις που έγιναν ε, ότι είναι υπερβολικές ε, οι δηλώσεις μου για τους Ρωμά και άλλα θέματα δεν θα τις σχολιάσω καν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Ταβάρη, τον ευχαριστώ και για τις προτάσεις και για τις παρατηρήσεις. Συμφωνώ με τις προτάσεις του και μάλιστα είπα ότι θα σας μοιράσω ένα έγγραφο λεπτομεριακό για την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Εκεί θα αναφέρω τις παρατηρήσεις με κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων αρμόδιων φορέων για την κατάσταση στα κράτη-μέλη και θα συνεργαστούμε όλοι μαζί στα θέματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, συναντήθηκα με εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και όπως είπατε κύριε Ταβάρες, μπορούμε να συνεργαστούμε κάλλιστα αποφεύγοντας φυσικά την επικάλυψη, κάνοντας οικονομίες μεγέθους και αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εκχωρήσουμε αρμοδιότητες μας, γιατί έχουμε το ρόλο μας, τις ιδιαιτερότητες και τις ευθύνες μας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι εταίρος που δεν τον ε, αξιοποιούμε παρκώς, αλλά είναι προνομιακός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν θα του θα το αναθέσουμε να μας υποκαταστήσει. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή της Κομεχάκης, φυσικά περιμένω την πρόταση και του Προέδρου και τη δική σας. Κυρία Τσίπελ, σας ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται από μια πρόσφατη δημοσκόπηση, ε, είναι σημαντικό αυτό το θέμα και καλό θα είναι να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Κροάτη συνάδελφο και μάλιστα η παρέμβαση του δείχνει το ενδιαφέρον του για αυτό το θέμα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και φυσικά θα πρέπει να εμπνευστούμε από το παρελθόν και από τις ε, εμπειρίες που είχαμε από τον φασισμό, τον ναζισμό, τον απολυταρχισμό, τον κομμουνισμό για να ενισχύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Ευρώπη και σε όλα τα κράτη-μέλη, τα παλιά και τα νέα. Γιατί διαπιστώνεται ότι ε, εκεί που μιλώ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, διαπιστώνεται ότι οι ίδιες παραβιάσεις έχουμε στις 15 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παλιές, ε, τις ίδιες παραβιάσεις σχεδόν έχουμε και στις καινούριε. Είναι σημαντικό λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά. Αυτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά συνοπτικός, αλλά παρόλα αυτά απάντησα. Ευχαριστούμε κύριε Μισελ. Προτείνω το εξή. Αυτό ήταν το σημείο που είχαμε ακριβώς πριν την ψηφοφορία που είναι προγραμματισμένη για τις 10.30. Ε, ήθιστε τα μέλη να περιμένουν ακριβώς την ώρα της ψηφοφορίας. Οπότε ας κάνουμε διάλειμμα για μισή ώρα και στις 10.30 θα ψηφίσουμε ώστε να γίνουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που είναι προγραμματισμένες για εκείνη την ώρα. Μου είπαν μόλις ότι ο κύριος Μούλτερ έχει τη γενέθλιά του σήμερα, οπότε χρόνια σας πολλά κύριε Μούλτερ. So, in half an hour we'll be having the vote. Σε μισή ώρα λοιπόν οι ψηφοφορίες.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

πολύ δυνατό να ότι με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 έρευνα στις λατρεύω, μου είναι έρευνα τώρα. Άλλο, κάτι μου μας πες άκρο, σαν τέλος. Да. Да. Да,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

Your colleagues? Your colleagues? Dear colleagues? Colleagues, thank you for your attendance. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ θερμά για την προσέλευση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 και είμαστε όλοι πολύ ακριβείς. 10 και 30 είχαμε προγραμματίσει την ψηφοφορία και είμαστε όλοι παρόντες. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέπειά σας. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Πρώτο θέμα, το σημείο 6 κατάλογος τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υπόχρηση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και κατάλογος τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Then, point number seven will be concerning the uh, flow. Και το σημείο 7 που αφορά την ε, ροή μεταναστών μετά τη σύραξη στη Συρία. έκθεση της κυρίας Μαρία Γκαμπριέλ πρώτα. Αλλά πριν την έναξη ψηφοφορίας, ζήτησε το λόγο η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ τώρα σε όλους τους συναδέλφους για να ζητήσω αναβολή της ψηφοφορίας. Ε, και αυτό γιατί στο, όνομα της διαφάνειας. Για αυτή την υπόθεση από την αρχή είχαμε εξαιρετική συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητέ Τους ευχαριστώ γι' αυτό. Έχουμε επίσης μια διαδικασία που ακολουθούμε. Θα ήθελα να θυμίσω το παιχνίδι αυτό Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη λήψη απόφαση σε ένα θέμα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο και πιστεύω πως εδώ ε, φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει, λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε ε, τις διαδικασίες. Είναι ένα μήνυμα διαφάνειας και διαλόγου. Ζητώ λοιπόν αναβολή της ψήφου διότι είχαμε προφορικές τροπολογίες που κατετέθησαν που αναφέρονται σε χώρες στις οποίες δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά που είναι απαραίτητο στο Κοινοβούλιο να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουμε να λάβουμε απόφαση εν γνώση όλων των στοιχείων. Γι' αυτό και ζητώντας την αναβολή της ψήφου έχω μία πρόταση να ζητήσουμε ε, ε, ε, ευγενικά να στείλουμε μια προταση να ζητησουμε ευγενικα να στειλουμε μια επιστελή στο όνομά σας στις τρεις χώρες που από ό,τι φαίνεται έχουν εδώ πλειοψηφία στο πλαίσιο της Επιτροπής μας, δηλαδή τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Περού και την Κολομβία, ώστε να μπορούμε να έχουμε από πλευρά τους, από τους πληροφορίες για το κατά πόσο είναι έτοιμες. Γιατί αυτά τα κράτη ζητούν σήμερα επί τη βάση κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται. Εάν όλα έχουμε τις πληροφορίες αυτές της διάθεσή μας, θα μπορούμε να λάβουμε απόφαση εν γνώση των ε, στοιχείων αν είμαστε υπέρ κατά μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να το κάνουμε σεβόμενη την διαδικασία, σεβόμενη τι αξίε διαφάνεια και διαλόγου και θα μα επιτρέψει ω Ευρωκοινοβούλιο να στείλουμε ένα μήνυμα και στα υπόλοιπα ε, θεσμικά όργανα αλλά και στου Ευρωπαίους πολίτες γιατί πρώτη φορά συμμετέχει σε λήψη, σε, ε, αλλά είναι και το θεσμικό όργανο που μεριμνεί ώστε όλα να γίνουν με σωστό τρόπο, με σεβασμό των κανόνων και με πλήρη διαφάνεια. Νομίζω πως τα είπα όλα και αφήνω την απόφαση φυσικά σε όλους μας. Είναι μια πρόταση που υποβάλλω στους συναδέλφους γνωρίζοντας εις βάθος την υπόθεση. Έχω την εντύπωση πως μπορούμε να λάβουμε μια αναπόφαση στο όνομα της διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαμπριέλ. Το μήνυμα ελήφθη. Ζήτησαν το λόγο όμως ε, συνάδελφοι. Ξεκινούμε από την κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ως σκιώδης ηγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να ευχαριστήσω την κυρία Γκαμπριέλ για τις προσπάθειές της και να συμφωνήσω με την πρότασή της για αναβολή της ψηφοφορίας ε, για δύο εβδομάδες γιατί μας ε, έδωσε πολύ βάσιμα επιχειρήματα για το αίτημα αυτό και μάλιστα λίγες ε, ώρες πριν την έναρξη ψηφοφορίας ε, έχουμε υποστεί πολλές πιέσεις ε, από πολλές χώρες για να προσθεθούν στον θετικό κατάλογο για το καθεστώς απαλλαγή θεωρήσεων. Πολλά μάτια είναι στραμμένα πάνω μας. Εξετάζουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να διερευνήσουμε την κατάσταση και να ζητήσουμε περισσότερα τεκμήρια χάρη διαφάνειας, όπως σας είπα. Και θα ήθελα να να σταθώ στο πλευρό ανεπιφύλακτα της εισηγήτριας. Είχαμε πολλές τροπολογίες τελευταία στιγμή και συζητούμε κάτι που θα μπορούσαν κάποιοι να μας κατηγορήσουν ότι παραβιάζουμε διαδικασίες. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Είναι τεράστια ευθύνη μας και δεν θα, θα ήθελα το αποτέλεσμα των σημερινών συζητήσεων να είναι σε βάρο ή να απογοητεύσει του πολίτε. Δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσει χωρί προηγούμενη εκτίμηση, αξιολόγηση τη κατάστασης και προηγούμενη σοβαρή συζήτηση. Και άλλοι σκιώδει ηγητές ζήτησαν το λόγο. Κύριε Λουμισέλ και σα σκιώδει είστε ή όχι. Κύριε Μισελ είστε σκιώδει. Μάλιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά τρέφω μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό προς τη Μαρία Γκαμπριέλ για το έργο της. Και φυσικά αντιλαμβάνομαι την επιχειρηματολογία της, αλλά δεν καταλαβαίνω την διαδικασία που μας προτείνει. Προτείνει αναβολή για δύο εβδομάδες. Διανοείστε δηλαδή ότι μέσα σε 15 μέρες θα στείλουμε την επιστολή και θα λάβουμε εγκαίρως τις εξηγήσει από τις 10 χώρες. Ε, κατά πάσα πιθανότητα θα αναβληθεί επαόριστον αυτή η ψηφοφορία. Τουλάχιστον θα προλάσουμε να ψηφίσουμε τρεχούς της κοινοβουλευτική θητείας. Το θέμα όμως είναι κατεπήγον. Και θεωρώ αξιολείπητο ότι οι 16 νησιωτικές χώρες ΑΚΕ που ήταν τελικά οι ενδιαφερόμενε χώρες ε, από την αρχή. Γιατί για αυτές τις 16 χώρες ε, ξεκίνησε η διαδικασία. Κρίμα είναι να, να γίνουν όμοιροι αυτής της αναβολής εξαιτία του λόμπι και της πίεσης που αναπτύχθηκε στη συνέχεια. Βέβαια, μου είπα ότι οι τρεις τροπολογίες, οι πιο επιμέχες και προβληματικές, ε, έχουν αποσυρθεί, ελπίζω. Οπότε έχουμε τελικά κάποιες χώρες που φαίνεται ότι χρήζουν ε, μεγάλης υποστήριξης. Γιατί λοιπόν, αφού μπορούμε να προχωρήσουμε και να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα για πολλές χώρες, γιατί να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Θα συμφωνούσαμε με την αναβολή εφόσον δεν είχαν αποσυρθεί οι τρεις επίμαχες τροπολογίες. Και όταν μου λέτε θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε την απόφαση όντας ενημερωμένοι και έχοντας γνώση της κατάστασης. Ναι, έχοντας γνώση της κατάστασης. Αλλά δεν μπορείτε να με πείσετε ότι οι κατατοπισμένοι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ και που ήδη έχουν εκφέρει τη γνώμη τους δεν ξέρουν από τώρα αν οι ελόγω χώρες είναι σε θέση να τύχουν απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων ή όχι. Θέλετε να πιστώ ότι μέσα σε 15 μέρες θα συγκεντρώσουμε ε, κριτήρια που θα τροποποιήσουν την ήδη κρατούσα θέση υποστήριξης ε, υπέρ των χωρών. Πολύ αφεβάλλω. Κύριε Κίρκοπ, προσοχή Λίγο χρόνο έχουμε, γιατί έχουμε μόνο μισή ώρα για την ψηφοφορία. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα τελευταία σχόλια. Εγώ διαπίστωσα από τον κατάλογο ψηφοφορίας με ιδιαίτερη χαρά ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα με τις προφορικές τραπολογίες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ε, να πιστεύουμε ότι θα μειωθεί στις επόμενες εβδομάδες ο κατάλογος των ε, χωρών. Μάλλον θα διευρυθεί. Να μην ε, γίνουμε όμως ξαφνικά ξεφραγομπέλοι και να υποβάλουν αθρώδεις υποψηφιότητες τους σε όλο και περισσότερες χώρες. Εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα, βλέπω κανένα δύο χώρες που είναι ε, επικρατέστερες. Αλλά Ούτω ή άλλως για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμπειράτα έχουμε εδώ και δύο χρόνια εντατικέ συζητήσει και διαπραγματεύσει. Και νομίζω ότι είναι θέμα σοβαρότητα απέναντι στη χώρα αυτή και σοβαρότητα δική μα και ανάληψη ευθύνη τη επιτροπή Να λάβουμε τι αποφάσει με βάση του κανόνε και με βάση το έργο που έχει γίνει ήδη και την προεργασία που έχει γίνει ήδη. Κατανοώ τα επιχειρήματα της ηγήτριας, αλλά αν δεν λάβετε εσείς την απόφαση ότι ε, δεν θα υπάρξουν αλλαγές ε, για τις υποψηφιότητες και δεν θα προσθεθούν υποψηφιότητες στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι που δεν είστε καν σε θέση να τις κάνετε, δεν θα ήμουν υπέρ της αναβολής, γιατί έτσι ίσως ε, βρεθούν σε δύσκολη θέση και οι δύο-τρεις υποψηφιότητες που ήδη πληρούν τις προϋποθέσεις. Είναι κρίμα να πληγούν οι χώρες αυτές. Η κυρία Στάνοκα, είμαι υπέρ της αναβολής γιατί πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα και δεν μπορούμε τελευταία στιγμή να εξετάζουμε προφορικές τροπολογίες λίγο πριν την ψηφοφορία. Θέλουμε συνεδρίαση των συντονιστών, των σχεδόν εισηγητών, συγγνώμη, για να δούμε σε τι θέση βρισκόμαστε και να εξετάσουμε σοβαρά την κατάσταση. Γιατί Έχουμε δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι η αναβολή χρειάζεται και μάλιστα όχι 15 ημερή, αλλά ενός μηνός. Κυρία Ένστ, ναι. να σας πω, ε, δεν είπαμε ότι θα καταργήσουμε, ότι θα το διαγράψουμε την ψηφοφορία, την ακυρώσουμε. Είπαμε για αναβολή και εμείς ε, συμφωνούμε σε αυτό υπάρχουν ορισμένοι αντιπρόσωποι κυβερνήσεων οι οποίοι ζήτησαν να μας συναντήσουν και ε, να μας παρουσιάσουν ε, ορισμένα στοιχεία και πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά και η Τάνια ε, μίλησε πράγματι σωστά. Δεν ζητήσαμε διαγραφή της ψηφοφορίας. Ζητήσαμε μόνο μία αναβολή. Χρειαζόμαστε περισσότερες, ψηφοφορίες έτσι ώστε να μπορέ... ε, περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε σωστά. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πω πολλά, πάντως το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι η έκφραση της ε, αναγνώρισης και της ευγνωμοσύνης μου προς την εισηγήτρια για το έργο της. Η κυρία Γκαμπριέλ που άλλωστε ανήκει και στην πολιτική οικογένεια και ξέρω καλά τι λέω. Όπως ξέρετε ήμουν κι εγώ τρεις φορές ηγητής ε, του κανονισμού 539-2001 και γνωρίζω τις δυσκολίες που έχουμε διοργανικά ε, για την διεκπαιρέωση της έκθεσης αυτής. Δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια να συμφωνούμε όλοι, ακόμη και εντός της ίδιας πολιτικής ομάδας και είναι υγιής η διαφωνία και η διάσταση απόψεων. Αλλά θα ήθελα πολιτισμένα, στοργικά αλλά και ταυτόχρονα κατηγορηματικά να εκφράσω τη διαφωνία μου με την πρόταση αναβολής. Και θα σας εξηγήσω για ποιους λόγους διαφωνώ. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί μπορώ να καταρρύψω το επιχείρημα της διαφάνειας. Ο κανονισμός είναι διαφανής και ο κανονισμός επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα που χρησιμοποιούμε. Επιτρέπει τη δυνατότητα άσκησης προφορικής τροπολογίας. Ως εκ τούτου, η διαφάνεια δεν είναι ασύμβατη με τον, ε, με τον κανονισμό. Αλλιώς δεν θα είχαμε αυτό τον κανονισμό που διέπει την πολιτική μας δράση. Άρα δεν ευσταθεί το επιχείρημα της διαφάνειας ως λόγος αναβολής. Δεύτερος λόγος. Δηλαδή μέσα σε 15 μέρες θα αποκατασταθεί η διαφάνεια, θα ενισχυθεί η διαφάνεια. Νομίζω ότι μερικοί ε, δεν το γνωρίζουν. Σας ενημερώνω όμως ότι η Κολομβία και το Περού έχουν ε, ε, καταθέσει τεχνικό δελτίο το οποίο έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί αναφέρονται με λεπτομέρεια τα διάφορα στοιχεία αξιολόγησης ε, που στοιχειοθετούν έγκριση ή απόρριψη του αιτήματο των δύο χωρών. Μάλιστα, ε, εμείς υποστηρίζουμε την ένταξη των χωρών με τον πρόεδρο Λόπες Αγγιλάρη και με την κυρία Ρενάτε Βέμπερ. Ούτως ή άλλως, αυτά τα σημεία καλύπτονται και από την εμπορική συμφωνία. Δεν μπορούσαμε να συνάψουμε εμπορική συμφωνία με την Κολοβία και το Περού, αν προηγουμένω δεν είχαν εκπληρωθεί αυτέ οι υποχρεώσει αμοιβαιότητα για την τήρηση των συγκεκριμένων σημείων. Για παράδειγμα, ανθρώπινα δικαιώματα και επίση σημαντική ασφάλεια των θεσμών της Κολομβίας και του Περού και η, η μεγάλη ποιότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων Ήδη έχουν βιομετρικά διαβατήρια οι δύο χώρες. Επίσης ε, ισχύει η αμοιβαιότητα. Δηλαδή, εγώ σε απαλλάσσω από υποχρέωση υποχρεώσεις και εμείς σε απαλλάσσουμε 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης και οι δύο χώρες ε, έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης στην ε, Αμερικανική Ήπειρο, στην Νότια Αμερική μάλλον. Όπως ξέρετε, Έχουμε πολύ περισσότερους Ευρωπαίους στις δύο αυτές χώρες από ότι περουάνου και Κολομβιανού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, εργασιακές ε, και εμπορικές σχέσεις. Άλλα επιχειρήματα που στοιχειοθετούν ε, την έγκριση αυτών των χωρών. Επίσης, το θέμα της ασφάλειας. Ένα θέμα που γνωρίζω πολύ καλά. Η ασφάλεια είναι ένα εχέγγυο αυτών των δύο χωρών, που ναι μεν έχουν προβλήματα, αλλά μην ξεχνάτε το εξής. Οι κυβερνήσεις και του Περού και της Κολομβίας έχουν αναλάβει δέσμευση για προσήλωση στην ασφάλεια. Και μάλιστα είναι αντικειμενική και απτή πια η δέσμευση που έχουν αναλάβει αυτές οι δύο χώρες υπέρ της ασφάλειας. Για όλους αυτούς τους λόγους και μια σειρά άλλων που δεν μπορώ να τους απαριθμίσω τώρα γιατί θα χρειαζόμουν πολλές ώρες, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην δεχτείτε το αίτημα της συγγήτριας Γαμπριέλ για αναβολή. Πρόεδρος, προτάθηκε αναβολή της ψηφοφορίας. Με βάση τον κανονισμό, όπως ισχύει και στην Ολομέλεια, όταν προτείνεται αναβολή της ψηφοφορίας από τον εισηγητή, μπορούμε να ακούσουμε ένα επιχείρημα υπέρ, ένα επιχείρημα κατά. Ακούσαμε ε, τις ε, απόψεις υπέρ. Ζητήθηκε και από την κυρία Τσίπελ ο λόγος, θα της τον δώσω και μετά θα ψηφίσουμε επί της αναβολής. Κυρία Τσίπελ, παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Πιστεύω πως ε, δεν είναι σωστό τώρα να διεξάγουμε μια συζήτηση σε βάθος για τα επιμέρους ε, κράτη. Τα κράτη αυτά έχουν παρουσιάσει τα επιχειρηματά τους, έχουν ήδη διεξαχθεί οι διεξοδικές συζητήσεις και πιστεύω πως ε, μια αναβολή δεν είναι και τόσο σωστή. Πιστεύω πως οι συνάδελφοι εδώ έχουν όφελος να εξετάσουν εάν πρέπει να αποσυρθούν ή όχι οι προφορικές τροπολογίες, ανεξάρτητα με την ε, συνέχεια. Είναι μια ε, εξέλιξη που έγινε τελευταία στιγμή, ούτε χθε ούτε προχθέ. Μετά από την ε, συνεδρίαση της πολιτικής μας ομάδας, χθε υποβλήθηκαν τροπολογίε και πιστεύω πως αυτό διακυβεύει την σοβαρότητα των συναδέλφων. Πιστεύω πως αυτή η διαδικασία και η τόσο τελευταία στιγμή είναι ακατάλληλη και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι καλό να αναβληθεί η ψηφοφορία έτσι ώστε να συζητήσουμε μεταξύ μας επί της διαδικασίας και βέβαια σχετικά με το περιεχόμενο και τις χώρες που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Προφανώς υπάρχει διχασμός της απόψεις Έχουμε την πρόταση της εισηγήτριας. Υπέρ της αναβολής και έχουμε και απόψεις κατά της αναβολής. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για να δούμε αν θα αναβληθεί η ψηφοφορία ή όχι. Αυτό ψηφίζουμε τώρα. Έχετε να ρωτήσετε κάτι επί του διαδικαστικού. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ε, ζητώ διευκρινήσεις σχετικά με τρεις προφορικές τροπολογίες. Τρεις προφορικές τροπολογίες που υπέβαλε έχουν αποσυρθεί. Ήδη ο κύριος Λουί Μισελ το ανέφερε, αλλά θα ήθελα να το ακούσω και από εσάς, ενώπιον μας. Ναι. Οι τροπολογίες 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 έχουν αποσυρθεί. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν αυτές τις τροπολογίες. Τώρα ψηφίζουμε για την αναβολή της ψηφοφορίας. Όσοι είναι υπέρ της αναβολής θα ψηφίσουν ναι, όσοι είναι κατά θα πρέπει να ψηφίσουν όχι. Ψηφίζουμε τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Το Άλικα έχει μία ψήφο παραπάνω. Για να δούμε λοιπόν. Πέρας. 32 ψήφοι υπέρ της αναβολής, 24 ψήφοι κατά. Αναβάλλεται λοιπόν η ψηφοφορία. Τώρα ψηφίζουμε για τη Συρία. Συρία λοιπόν.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 Κυρία Βίξτρομ, έχετε να πείτε κάτι επί του διαδικαστικού. Πρόεδρε, προτείνω να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για τη Συρία. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα ψηφοφορία για τη Συρία. Καθίστε παρακαλώ, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, κάντε το σιωπηλά. Κυρία Βίξτρομ. Ναι συζητούμε επί της διαδικασίας όταν έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ψηφοφορία για τη Συρία και βλέπω πως πολλοί φεύγουν από την αίθουσα και το θεωρώ απαράδεκτο. Ας προχωρήσουμε αμέσως λοιπόν στην ψηφοφορία. Αυτό θα κάνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Έπρεπε να ψηφίσουμε για αναβολή και τώρα θα ψηφίσουμε για τη Συρία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Τι θέλετε να... εσείς επί του διαδικαστικού. Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα είναι συνενετικό. Υπάρχει όμως μια δημοσιονομική δυσκολία γιατί έχει περικοπεί ο προϋπολογισμός. Τα κονδύλια έχουν μειωθεί. Γιατί μερικές ομάδες στάχθηκαν κατά της αύξησης των κονδύλιων για τους ε, μετανάστες και είναι ε, αντίφαση. Να υπάρχει συνένεση για το ψήφισμα, αλλά όχι συνένεση για τον προπολογισμό. Καλό το ψήφισμα, αλλά ίσως είναι τελικά απλώς ωραία λόγια. Ξύλινη γλώσσα. Vote. Ψηφίζουμε τώρα λοιπόν για τη Συρία. Τροπολογίες. Τροπολογία 1. Υπέρ. Ωραία. Unblock. Συμφωνείτε? Ωραία, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτονται οι 7 τροπολογίες και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 43 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλέης, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε την κάθε τροπολογία ξεχωριστά δεν θα μας έπαιρνε ώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις ψηφίσαμε unblock. Και δεν πιστεύω πως αυτό είναι αδικαιολόγητο. Μάλιστα, το σημειώσαμε. Υπήρξε η πρόταση από τους συντονιστές να ψηφίσουμε τις τροπολογίες unblock και όλοι συμφώνησαν αμέσως. Αυτό έγινε. Τοποθετηθήκατε, μάλιστα.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 8 το πρωτόκολλο σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων ε, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή η Χρυσή Αυγή. Η συγγήτρια είναι η κυρία Βερονίκα Ματιού Ουγιόν, αλλά κολλείεται από ό,τι ξέρω. Οπότε θα την αντικαταστήσει ο κύριος Άξελ Βος. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης και θα ακούσουμε και τους κοιόδης ηγητές. Αυτά. Κύριε Φως, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσω εκ μέρους της Βερονίκ Ματιέ και θα σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης. Δυστυχώς η κυρία Ματιέ απουσιάζει, μου ζήτησε όμως να την εκπροσωπήσω. Ε, καταρχάς η Βερονίκ Ματιέ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους κοιόδης εισηγητές για την καλή συνεργασία και τη στήριξη που τη έδωσαν. Ε, το θέμα είναι το πρωτόκολλο για την ε, παράνομη μετα... ε, κατασκευή, μεταφορά ε, πυροβόλων όπλων εκρηκτικών και πυρομαχικών. Το θέμα λοιπόν είναι η παράνομη κατασκευή και η πρόληψη, καταστολή και δίωξη της ε, παρανομής κατασκευής. Είναι συμπληρωματικό πρωτόκολλο στο, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το ε, διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν επίσης δύο συμπληρωματικά πρωτόκολλα, το ένα για την παράνομη μεταφορά μεταναστών και το άλλο για την πρόληψη καταστολή και δίωξη ευπορίας προσώπων, τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το πρωτόκολλο το 2000, ε, υπέγραψε το πρωτόκολλο το 2002 και δεσμεύτηκε για την έγκρισή του και από τη στιγμή μάλιστα που θα, από τη στιγμή που θα εναρμονιστεί με την κοινοτική νομοθεσία. Υπάρχει μία ε, ενοποιημένη διαδικασία όσον αφορά την ε, παράνομη κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων, όπλων, εξαρτημάτων, μερών και πυρομαχικών και με την οδηγία 51-2008 ε, εισήχθησαν νέες διατάξεις. Ο κανονισμός 258 του 2012 ως ε, συμπληρωματικός του άρθρου 10 δημιουργεί ένα πλαίσιο για την ε, έγκριση και τις απαιτήσει ε, αδειοδότησης όσον αφορά την εισαγωγή, εξαγωγική διαμετακόμιση και ελέγχους. Η συγγήτρια μέσω της έγκρισης του πρωτοκόλλου θεωρεί πως όλα τα κράτη-μέλη θα θα δεσμευτούν ε, νομικά πλέον για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου να τονίσω τέλος ότι το παράνομο εμπόριο των πυροβόλων όπλων έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει η τελευταία έκθεση της Ευρωπόλ, της, ε, ΣΟΚ, της ομάδας ΕΣΟΚΤΑ, η οποία δείχνει ότι το εμπόριο όπλων έχει γίνει κυρία πηγή εισοδήματος ε, για εγκληματικές οργανώσεις σε 18 χώρες έχουν αναφερθεί 39 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες ε, ασχολούνται με το εμπόριο όπλων ως κύρια δραστηριότητα και ως ε, παράλληλη δραστηριότητα άλλες 14 εγκληματικές οργανώσεις. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι ως εισηγητής χαίρομαι πάρα πολύ που ο αγώνας για την ε, καταπολέμηση και καταστολή του και δίωξη του εμπόριου όπλων είναι μία από τις προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα πλαίσια της στρατηγικής για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν νομικές ε, διατάξεις του πρωτοκόλλου οι οποίες ενισχύονται από αυτά τα στοιχεία όπως για παράδειγμα η σήμανση και η τήρηση λεπτομερών αρχείων για τα πυροβόλα όπλα και για τις ε, άδειε. Η συγκήτρια επίσης θέλει να τονίσει την, ε, σημασία, την, ε, την μεγάλη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 12 του πρωτοκόλλου, διότι η διεγκληματικότητα δεν γνωρίζει σύνορα και το εμπόριο όπλων θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μόνο όταν βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και μόνο όταν ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι καλύτερα δικτυωμένα και συνδεδεμένα στη συνεργασία τους από ότι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις. Φυσικά χρειάζονται ε, τα κατάλληλα μέσα για την καταπολέμηση του παράνομου εμπόριου όπλων. Υπάρχουν πάρα πολλά παράνομα πυροβόλα όπλα τα οποία προέρχονται από τα Βαλκάνια και την Ρωσία και διοχετεύονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα καλά σνικόφα για παράδειγμα. Και η εισηγήτρια θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν ανταλλάσσουν αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η απειλή αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο ε, μέρος αυτών των όπλων προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό ζητείται από τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βελτιωθεί το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρωπόλης, το οποίο ε, παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 20 διαφορετικών ε, στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογούνται και θα εξετάζονται ξεχωριστά. Και η συγγήτρια επίσης χαιρετίζει τη σύσταση για δημιουργία μιας κεντρικής θέσης ε, στα πλαίσια της Ευρωπόλ για την η καταπολέμηση του παράνομου εμπόριου όπλων, η οποία κεντρική θέση επίσης θα αναλάβει ε, αυτό το πολύ σημαντικό έργο και θα πρέπει να τύχει σημαντικής και στρατηγικής στήριξης. Από τη στιγμή που εναρμονιστεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να εγκριθεί και το ε, πρωτόκολλο για το για την παράνομη κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων όπλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρωτόκολλο, όπως είπα, και μας δίνει τη δυνατότητα η έγκρισή του ε, για την καταστολή και δίωξη αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες ε, έχουν πάρα πολύ μεγάλο εύρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η συγγήτρια λοιπόν είναι υπέρ, σαφέστατα υπέρ της ε, έγκρισης του πρωτοκόλλου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Έχουμε εδώ τον Κλοντ Μωράης που είναι πρόθυμος να παρέμβει. Στη συζήτηση. Ευχαριστώ, Χουάν. Εγώ ήθελα πολύ σύντομα να πω ότι ο κύριος Βος έκανε μια πολύ εμπεριστατωμένη εισήγηση για τις προθέσεις της κυρίας Ματιέ για αυτή την έκθεση. Και ως κοιόδης των σοσιαλιστών θέλω να εκφράσω την πλήρη μας στήριξη για τη θέση της εισηγήτριας. Φυσικά, επειδή την υποστηρίζουμε πλήρως, δεν σκοπεύουμε να υποβάλουμε τροπολογίες, γιατί θέλουμε γρήγορα να λυθεί ε, αυτό το θέμα, να ψηφιστεί γρήγορα αυτό το πρωτόκολλο του ΟΗΕ. γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα και ε, <clears throat> συμφωνούμε όλοι οι σκιώδες γι' αυτό, όπως φάνηκε και από τις συνεδριάσεις. Δεν ε, έχω πολλά να πω μετά από την εισήγηση του κυρίου Βος. Πολύ σημαντικό το θέμα για μας. Το... Να... Η παράνομη κατασκευή αλλά και το εμπόριο είναι θέμα που πρέπει γρήγορα να λυθεί. Συμφωνούμε όλοι και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει γρήγορα συμφωνία σε ολόκληρο το ΣΕΜ. Ευχαριστώ τον κύριο Βόζ για αυτή την εμπεριστατωμένη εισήγηση εξ ονόματος τη κύρια Ματιέ και ελπίζω ότι θα ε, ολοκληρωθεί γρήγορα η εξέταση του θέματος. Ευχαριστώ. Κύριε Μωράης, δεν έχω κανέναν άλλον που να θέλει να παρέμβει. Κομισιόν, το Συμβούλιο θέλει να προβεί σε κάποια δήλωση. Όχι. Όχι. Ούτε η Κομισιόν, ούτε το Συμβούλιο. Θέλετε κάτι να προσθέσετε. Όχι. Κύριε Βόζ, εσείς που αντιπροσωπεύετε την εισηγήτριά μας την κυρία Ματιέρ, όχι. Μάλιστα. Αυτό θέλαμε λοιπόν, να εξετάσουμε την, ε, το σχέδιο έκθεση και να θεσπίσουμε ημερομηνία για υποβολή τροπολογιών το μεσημέρι, στις 12. Εντάξει. Αυτά λοιπόν, γιατί όπως είπα, η συνεδρία των συντονιστών έχει αναβληθεί και δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε μέχρι τις 3 όπου θα συνεδριάσουμε εκ νέου. Γεια σας.